Αγαπητοί βουλευτές, με το άνοιγμα της νέας αυτής συνόδου, για άλλη μια φορά, είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε αθώα θύματα της ε, οργής του, της διεθνής τρομοκρατίας. Εξ όλων καταδικάζω στέναρα αυτές τις πράξεις απάνθρωπης βίας και εκφράζω την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής βίας της Βαρκελόνης και της φιλανδικής πόλης της Τούρκ και του Καμπρίλ. Βεβαίως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες σε μη ευρωπαϊκές χώρες που γνωρίζουν αυτή τη βαρβαρότητα. Σήμερα στις 11 ε, Σεπτεμβρίου διανύουμε την 16η χρονιά μετά την τρομοκρατική αυτή ενέργεια της 11 η Σεπτεμβρίου το 2001 και πρέπει να καταδικάσουμε από κοινού την τρομοκρατία και να θωρακιστούμε κατά καλύτερο τρόπο έναντι της τρομοκρατίας. Είμαστε υπερήφανοι για τη ζωή μας για τις ελευθερίες μας και για τη δημοκρατία μας που θα υπερασπιστούμε, χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκύψουμε το κεφάλι μπροστά στην τρομοκρατία. Δυστυχώς όμως σήμερα θα πρέπει να τιμήσουμε άλλα αθώα θύματα που έχασαν τη ζωή τους μετά από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν μέχρι χτες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες της Καραϊβικής καθώς και της ΗΠΑ. Υπενθυμίζω την ύπαρξη αυτών των αθώων θυμάτων και θα ήθελα να τηρήσουμε όλοι ενός λεπτού σιγή. Ο κύριος Ντάντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χτες το βράδυ στο Λιβόρνο δυστυχώς σε λίγες ώρες ε, έπεσε τόσο νερό όσο τους τελευταίους οκτώ μήνες. Αυτό δημιούργησε οδήγησε μάλλον στην ύπαρξη έξι θυμάτων, μια ολόκληρη οικογένεια και υπάρχουν και δύο αγνοούμενοι. Εσείς υπενθυμίσατε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας και των φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα όμως να υπάρξει έμπρακτη αλληλεγγύη με συλληπιτήρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την πόλη του Λιβόρνο, διότι γνωρίζει μεγάλες ε, ζημιές που πρέπει να αντιμετωπιστούν και επίσης να μιλήσουμε και κατά των κλιματικών αλλαγών που έχουν οδηγήσει σε αυτά τα θλιβερά συμβάντα όπως αυτό στην δική μου περιφέρεια αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Θα ήθελα λοιπόν να αναλάβουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις κατά των κλιματικών αλλαγών. Κύριε Ντάντη, συμμερίζομαι τα λεγόμενά σας γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και τα γεγονότα εντός και εκτός Ευρώπης μας οθούν να οθήσουμε, να προωθήσουμε αυτά μας τα συμφέροντα. Ο κύριος Πιτέλα, μιλήσατε για τις τραγωδίες των τελευταίων ωρών, συμμερίζομαι τα λόγια σας και υπενθυμίζω τη δραματική τρομοκρατική ενέργεια κατά των δίδυμων πύργων. 44 χρόνια πριν, στις 11 Σεπτεμβρίου, στην Κάσα Ροσάδα, στο Σαντιάγο της Κιλής, σκοτώθηκε ένας μεγάλος δημοκράτης ηγέτης, ο μέγας σοσιαλιστής Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε ήμουνα 14 χρονών όταν άκουσα αυτό το νέο από το ραδιόφωνο. Τα λόγια του είναι, μου είναι εντυπωμένα. Είπε, μπορείτε να με σκοτώσετε αν θέλετε, αλλά ποτέ δεν θα σκοτώσετε τα ιδεώδη και τις αξίες μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας καθοδηγούν τα λόγια του Σαλβαδόρ Αγέντε, γιατί μπορούμε να καταδικάσουμε κάθε επίθεση κατά της ελευθερίας και της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πιο δυνατή Ευρώπη και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο κύριος Προύστ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτό το λεπτό σιγής, ε, ιδιαίτερα για τον ε, τυφώνα που έπληξε την Καραϊβική και ειδικά τον Άγιο Μαρτίνο και τον Άγιο Βαρθολομαίο. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα πράγματα. Και θα ήθελα να χαιρετήσω την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ υπό την αιγίδα του κυρίου Στυλιανίδη και από τις Βρυξέλλες και επιτόπου. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε αυτές τις προσπάθειες, γι' αυτό θα ήθελα να κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για μια στρατηγική αποκατάστασης και αναδιάρθρωσης. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και περίσκεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ορίσουμε νέα σενάρια και κινδύνους και να διαχειριστούμε τις κρίσεις πολύ καλύτερα υπέρ των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας και την ε, υπηρεσία πολιτικής ασφάλειας που υπάρχει στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Προύστ. Όπως είπατε πολύ σωστά, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ζητήσουν την εκκίνηση δράσης του Ταμείου Αλληλεγγύης. Νομίζω ότι η Γαλλική Δημοκρατία θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και θα ζητήσουμε ένα δις 200 εκατομμύρια για την ε, Ιταλία, την κεντρική Ιταλία που επλήγει από το μεγάλο σεισμό και όπως ξέρετε θα υπάρξει ταχεία ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αποσταλεί ένα μήνυμα απτής αλληλεγγύης προς τους ε, Γάλλους πολίτες που επλήγησαν από την ε, φυσική αυτή καταστροφή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ιταλίας, θα ψηφίσει εντάχει όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκκίνηση χρήσης κονδυλίων από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ο κύριος ε, Καρίν και μετά ο κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, σήμερα το πρωί διάβασα μία έκθεση που δημοσιεύτηκε στο ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους EU Citizens και εκεί αναφέρεται η κατάσταση που διαμορφώνεται. Η Βρετανική κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα ο αρμόδιος υπουργό ε, έχει επιληφθεί του θέματος και θα ήθελα το γραφείο σας να βοηθήσει την Βρετανική κυβέρνηση έτσι ώστε αυτό το θέμα να εξαφανιστεί για να μην υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση. Αυτό μου θυμίζει την εποχή όπου υπήρχαν πινακίδες που έλεγαν απαγορεύεται είσοδος σε σκυλιά και σε μαύρους. Απαράδεικτο. Και πλέον κύριε Πρόεδρε όσον αφορά ε, στην απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Μα τι είναι αυτό που κάνουμε τη στιγμή που ε, το βραβείο δίδεται σε ανθρώπους ε, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κατά του πνεύματος που χαρακτηρίζει το βραβείο. Πώς είναι δυνατόν να επιβραβεύουμε τέτοιου είδους καταστάσεις με την απονομή του βραβείου που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρεμβαίνει κανείς σε, σε αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί σχετικά με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ε, ε βεβαίως ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά όσων έχουν λάβει το βραβείο Σαχάροφ και να καταδικάσουμε τη συμπεριφορά τους εκ των υστέρων. Εν πάση περιπτώσει θα περιμένω και θα δω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο εκ των υστέρων να παρέμβουμε σε αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Κάρβερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα και να πω ότι πράγματι εκφράζουμε τα συλληπιτηριά μας για αυτά που διαδραματίστηκαν στις γαλλικές υπερπόντιες περιοχές. Ε, όμως ε, υπάρχει, υπάρχουν και άλλες καταστροφές, αυτές που έχει προκαλέσει ο κυκλώνας Ήρμα. Ε, πολλές ανεξάρτητες χώρες έχουν πληγεί, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφέρουμε όλες τις χώρες, είτε είναι, ανήκουν στη Βρετανία είτε στη Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πλήγησαν, γι' αυτό λοιπόν ας εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους γίνεται. Πρόεδρος, ε, κοίταξε, εγώ δεν έκανα καμία διαφοροποίηση. Εγώ είπα ένα λεπτό σιγής για όλους ε, για να τιμήσουμε ε, όλα τα θύματα στην ευρωπαϊκή επικράτεια αλλά και εκτός Ευρώπης θύματα τα οποία επλήγησαν από τις κλιματικές αλλαγές. Ε, το ίδιο και για την τρομοκρατία. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στα θύματα και όσον αφορά στο Ταμείο Λεγγύης νομίζω ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να λάβουν τις ε, σχετικές αποφάσεις. Ε, Χιμένες Μπεβερίλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω, ξέρω ότι υπενθυμίσατε όλα τα θύματα και όπως είπατε δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ θυμάτων, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα θύματα του σεισμού του Μεξικού με πάνω από 100 νεκρούς. Είναι μια χώρα εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε το Μεξικό και την κυβέρνησή του. Ευχαριστώ. Ως, ως ε, πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου, πολύ σωστά είπατε ότι ε, θα έπρεπε να αναφέρουμε και τα θύματα του σεισμού στο Μεξικό. Το εννοούσα αυτό όταν είπαμε να λεπτό και για όλες τις άλλες κατακλυσμιές καταστροφές και φαινόμενα που έχουν προκύψει. Λοιπόν, προχωράμε της εργασίας μας. Ε, συνεχίζουμε την Ολομέλεια που είχε διακοπεί τον Ιούλιο του 2017. Ε, Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Κατόπιν τούτου τα πρακτικά εγκρίθηκαν. Μετά από την